Uh, good morning, colleagues. Um, Καλημέρα σας. Θα αρχίσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις τότε εγκρίνεται. Για τις γλώσσες. Μόνο γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ζωηδικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβακικά, βουλγαρικά και ρουμανικά σήμερα η έγκριση των συστάσεων των συντονιστών τακ, τακ, τακ. πρέπει να σας πληροφορήσω ότι οι συντονιστές λόγω του περιορισμένου αριθμού των συνεδριάσεων που εγκρίθηκαν το 16 ζήτησαν δύο περισσότερα σμότ την 5η 14 Ιανουαρίου και την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο η δεύτερη. Δέχεστε αυτές τις συστάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε όλοι τις κάρτες σας. Αν κανείς δεν έχει, να το δηλώσει. Ωραία. Καλημέρα και σε όσους μόλις ήρθαν. Και μόλις κατάλαβαν ότι μιλάω, γιατί είναι, έχει κάποιο πρόβλημα το μικαρόφωνο. Δεν σας αρέσει η φωνή μου. Α, λέτε ότι μιλάω πιο δυνατά. Καλά, αυτό καλό είναι. Πιο δυνατά θα πει με περισσότερο κύρος, λοιπόν. Αφού έχουμε να κάνουμε με τόσο σημαντικό κανονισμό, είπα και εγώ να τα πω πιο δυνατά, τέλος πάντων. Αφού έχετε τις κάρτες σας, έχουμε τρεις ψηφοφορίες σήμερα. Να μείνετε και για την τρίτη, τρεις, τρεις. Πριν αρχίσουμε όμως, θα ήθελα να σας πω ότι μερικοί δεν θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα όπου θα γίνει η πληροφόρηση της Προεδρίας και τα λοιπά. Μερικοί ήδη το έχουν δηλώσει. Ήθελα λοιπόν να σας πω πολύ σύντομα ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πρωτοφανής αριθμός τριμερών διαλόγων που έχουν σχεδόν συμπληρωθεί ή έχουν συμπληρωθεί για την Επιτροπή μας και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτάς που πήραν μέρος τους Κιώδης και όλους τους υπόλοιπους Να ευχαριστήσω επίσης τα μέλη της ε, γραμματείας της ΛΥΜΠΕ διότι σας είπα ήταν μεγάλος ο φόρτος εργασίας και πρωτοφανής γιατί ήταν πιο μεγάλος ο αριθμός των θεμάτων μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Ιδίως εκείνους που δεν θα μπορέσουν να έρθουν στις τελικές μας συνεδριάσεις την επόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσει σε λίγο και η Προεδρία. Θα τους ευχαριστήσω αφού μιλήσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δηλαδή την έκθεση Albrecht. Η ψηφοφορία του κειμένου θα γίνει λοιπόν ηλεκτρονικά, είναι ονομαστική. Ο εισηγητής κύριος Άλμπρεχτ μήπως θέλει να μας πει τίποτε. Ορίστε. Make it uh, short, but I would also like to take the opportunity to uh, thank um, very much my negotiation team, the Shadows, who uh,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 Ας πούμε, ε, περάσαμε το θέμα του δικαιώματος να ξεχαστεί κανείς, κάτι που στην ουσία μας επέτρεψε να δώσουμε χώρα για μια νέα καινοτομία, για ίσους όρους ε, για τις εταιρείε ε, που θέλουν να μπουν στην ψηφιακή αγορά, η οποία με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται και αυτά τα δικαιώματα ε, τα προσπίσαμε με ισχυρές αρχές και κάτι τέτοιο ήταν από την δική μας πλευρά νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Uh, Ευχαριστώ, Γιάν. Ε, μια πολύ σημαντική παρέμβαση τώρα από την πλευρά της Προεδρίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω λίγα λόγια εκ μέρους ε, της ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου. Καταρχάς, ε, να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για αυτή τη μεταρρύθμιση στο σώμα, στην Επιτροπή σας, τον εισηγητή, τον κύριο Άλμπρεχτ, τον κύριο Λαγκριστίν για τη δουλειά του επίσης, του Σκιώδης και όλες τις ομάδες. Επίσης, ευχαριστώ όλη την ομάδα του, ε, τη διαπραγματευτική του Λουξεμβούργου και του συναδέλφου μου που δουλεύουν στις Βρυξέλλες. Οι τελευταίοι μήνες ήταν εντατικοί, όμως ε, το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο γιατί καταφέραμε να έχουμε μια καλή και δίκαιη συμβαστική λύση που θα είναι καλή για τους πολίτες της Ευρώπης ε, και τους επιχειρηματίες. Η ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου εχθέ ενημέρωσε την Κορεπέρ για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και το τελικό πακέτο. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν για την Προεδρία ότι η μέγιστη πλειοψηφία των κρατών μελών υποστηρίζει το τελικό πακέτο, τον κανονισμό και την οδηγία. Μετά τη δική σας ε, ψηφοφορία σήμερα θα επιστρέψουμε αύριο το απόγευμα στην Κορεπέρ και θα ζητήσουμε την επιβεβαίωση αυτού του συμβαστικού κειμένου από τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να έχουμε συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Η Προεδρία είναι πεπισμένη ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών θα επιβεβαιώσουν αυτή την έγκριση και ελπίζουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα υποστηρίξουν αυτή την ε, συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Θα κατευχαριστούμε. Τώρα αρχίζει η ψηφοφορία. Ονομαστικά. Άρχεται. συνάδελφοι έχουμε δύο παραπάνω από το ΕΛΚ okay, stay calm, um, just one now, Ένας τώρα παραπάνω. Ένας παραπάνω. Εντάξει τώρα. Ψήφισαν όλοι. Έληξε. Εγκρίνεται. 48-4 με τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επόμενη ψηφοφορία τώρα του κύριου Μάριου Λαουριστίν. Ο εισηγητής είναι λοιπόν ο κύριος Λαουριστίν. Μήπως κύριε Λαουριστίν μου θέλετε να πείτε τίποτα. Κυρία, κυρία. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου Να σας ευχαριστήσω για τους, να ευχαριστώ τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα. Είμαι καινούρια στο χώρο αυτό και είχα ένα κείμενο μπροστά μου το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί και χρειάστηκε να πάω προς την τελική ψηφοφορία. Έμαθα πάρα πολλά και από τον Τίμωθη και από τον Γιάννη και από τη Σοφή. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο ελπίζω θα μας οδηγήσει σε μια νέα κατάσταση με την επιβολή του νόμου στην Ευρώπη. Μιλάμε για την πρώτη εναρμόνιση του νομικού πλαισίου και ελπίζω πως εδώ θα αυξήσουμε το επίπεδο αλληλοκατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό στην ανταλλαγή πληροφοριών, πόσα προβλήματα είχαμε. Ελπίζω λοιπόν σε μια βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ διοκτικών αρχών στι χώρε μέλη, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικέ και να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ τη προστασία, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του ιδιωτικού χώρου, των ε, προσωπικών δεδομένων, που θα συνοδεύονται από μια παράλληλη ε, αποτελεσματική επιβολή του νόμου. Θέλουμε μια νέα εποχή ανταλλαγής πληροφοριών να ανατείλει και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο διαπιστώσαμε πως ε, σταδιακά τα κράτη-μέλη πλησίασαν τις θέσεις αλλήλων στην αρχή θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Προεδρία του Λουξεμβούργου γιατί έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να προσεγγίσουν ε, μια λύση για να πετύχουμε και την ε, τελική αυτή λύση. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη Ματίλδα, την Ελένη, το υπόλοιπο προσωπικό αντιμετωπίσαν τεράστιες πιέσεις τους τελευταίους μήνες, συνεχίζανε τη δουλειά τους νύχτα μέρα και Σαββατοκύριακα. Το ίδιο και για τους σκιώδεις, οι οποίοι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν ένα πολύ σκληρό χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω πως το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για τα κράτη-μέλη, για εμάς και για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη. Thank you very much, Mario. Ευχαριστώ πολύ Μάριο. Για την οδηγία αυτή λοιπόν θα ξεκινήσει η ψηφοφορία άρχεται. So, colleagues, um, for the EPP we have... Συν έναν από το ΕΛΚ. Σας παρακαλώ πολύ διορθώστε το. Um, if colleagues for the EPP just to correct... Συνάδελφοι από το ΕΛΚ, ακόμα είμαστε συνένα από την πλευρά σας. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 53 υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια για την εισηγήτρια. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μία ψηφοφορία έχει μείνει όχι τόσο μεγάλη ιστορική σημασία και θα ήθελα να, μου, να σας ζητήσω ε, συγγνώμη που την βάλαμε στο τέλος είναι για τα οχήματα και την κατάταξη στην Λετωνία ξεκινάμε λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία ναι εάν θέλετε συνάδελφοι είμαστε έτοιμοι λίγη ψηφοφορία ωραία εγκρίνεται ωραία έληξαν οι ψηφοφορίες για όσους δεν είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα, καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και για όσους θέλουν να πιούν ένα ποτήρι σαμπάνια, σας περιμένουμε στο μπαρ αμέσως έξω από την αίθουσα. Ξέρουμε πως είναι νωρίς, αλλά θέλαμε να σας προσφέρουμε ένα ποτήρι σαμπάνια.